Θα ήθελα δηλαδή να αποτίσω φόρο τιμή σε όλου εκείνου, στη δίδα μου τη βοηθό, αλλά και σε όλου του βοηθού μα και συνεργάτε μα που έχουν ε, τόσα πολλά προσφέρει στην προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακέβαν. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στι 12 το μεσημέρι. Και έτσι ε, αύριο αρχίζει 8.30 η συζήτηση μέχρι τις 2, μετά από τις 3 μέχρι τις 8 και από τις 9 έως τις 11 το βράδυ και ε, διακόπτουμε για σήμερα τη συνεδρίαση.